σημείο 19. Ο κανονισμός ο λεγόμενος για την πρόσβαση στην αγορά. Όπως ξέρετε, Είχαμε κάποιες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, φτάσαμε σε ένα συμβιβασμό, είμαστε στη δεύτερη ανάγνωση απαιτείται απλή πλειοψηφία. Ε, απόλυτη πλειοψηφία θα απαιτηθεί στην Ολομέλεια. Όπως ξέρετε, η αντιπροσωπεία του ΕΛΚ έχει ευελιξία στις ε, διαπραγματεύσεις και διαπραγματευόμαστε πάντα με βάση ε, μια βάση ad referendum. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πως τώρα πρέπει να επιβεβαιώσετε ή να μην επιβεβαιώσετε ε, αυτά τα οποία επιτύχαμε στις διαπραγματεύσεις μας με το ε, Συμβούλιο. Ας ψηφίσουμε λοιπόν. Συμβιβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Τα αποχές δεκτή. Θέλετε να το επαληθεύσουμε. Ε, έχετε το δικαίωμα βεβαίως. Να την επαληθεύσουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. υπάρχει ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Μια κάρτα πρέπει να βγει, ωραία. Κάποιοι λείπουν. Υπάρχει ακόμα ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. εξακολουθεί να υπάρχει ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Κάποιος από το ΕΛΚ πρέπει να βγάλει την κάρτα του. τώρα είναι εντάξει. Μάλιστα. Πέρας. Εγκρίνεται 19 υπέρ 4 ε, κατά 7 αποχές τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το σχέδιο σύστασης ψήφισμα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21, κατά, 21 υπέρ, 5 κατά, 4 εποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ 5 κατά 4 4 κατά 5 αποχές με συγχωρείτε συγχαρητήρια στην αντιπροσωπεία την διαπραγματευτική και τον εισηγητή επόμενο σημείο το 20 Πρόκειται πάλι για ένα νομοθετικό φάκελο με εισηγητή τον David Martin για να επανεισαχθεί η μια Βερμανία στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Υπάρχει μια τροπολογία. Υπαριθμών 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία του σχεδίου έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. 27 υπέρ, 2 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. υπέρ 2 κατά εγκρίνεται. Δεν υπάρχει αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Item 21. Σημείο 21. Κανονισμός ε, για την ε, χρηματοοικονομική ευθύνη που σχετίζεται με την εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων ε, σε εθνική συμφωνίες στις οποίε είναι συμβεβλημένο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν 7 συμβιβαστικέ τροπολογίες από 122 που ήταν αρχικά. Τον λόγο έχει ο εισηγητή για να μα εξηγήσει και τη θέση, να μας εξηγήσει τη διαδικασία και τη θέση του. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συναδέλφους, τους σκιώδησίτες και το προσωπικό. Θεωρώ πως κάναμε πολύ καλή δουλειά και καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Θεωρώ πως ε, με την έκθεση αυτή τελειώνουν ε, σχεδόν τρία χρόνια δουλειά μας στην ε, Επιτροπή για την προστασία ξένων επενδύσεων κάτι το οποίο αποτελεί συνέπεια των νέων αρμοδιοτήτων μας αρμοδιοτήτων μας έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας όμως Ε, φάνηκε στις συζητήσεις κάποια ζητήματα είναι ακόμα ανοιχτά πρώτα απ' όλα. Υπήρχε ζήτημα εσωτερικών διμερών επενδυτικών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ακόμα εκκρεμούσαν και δεν είχε ξεκαθαρίσει το ζήτημα από κανένα νόμο μέχρι στιγμής και θεωρώ πως υπήρχε μια άνηση μεταχείριση μεταξύ ε, Ευρωπαίων ε, επενδυτών. Οπότε έπρεπε να δούμε αυτό το ζήτημα με κάποιον τρόπο. Και μετά υπάρχει το πολύ σημαντικό ζήτημα της ίσης ε, μεταχείρισης των ε, Ευρωπαίων επενδυτών ε, σε σχέση με τους ξένους. Κάποιες χώρες όπως η ΕΠΑ έχουν τέτοιες λύσεις που εγγυώνται ίσου όρους ανταγωνισμού. Και θεωρώ πως με αυτά τα άλλα ζητήματα θα χρειαστεί ίσως να κάνουμε ίσως κάποια ακρόαση, κάποιο ψήφισμα για να επισημάνουμε τα προβλήματα τα οποία στην περίπτωσή μας θα πρέπει να λυθούν από την Επιτροπή. Να τονίσω επίσης πως ε, τα ζητήματα αυτά τα έθεσαν και κάποιες ε, πολιτικές ομάδες και συμφωνήσαμε πως ε, αυτή η περαιτέρω δουλειά της Κομισιόν θα οδηγήσει σε κάποια λύση. Οπότε γι' αυτό ζήτησα να επεξεργαστούμε περαιτέρω αυτά τα ζητήματα. Ε, για την ψηφοφορία. Μετά την ψηφοφορία θα, θα εξηγήσω την, την διαδικασία. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνω δύο παρατηρήσεις. Ε, με ενημερώσατε. Με ενημέρωσαν για το θετικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με τις άλλες ε, πολιτικές ομάδες και πρέπει να πω πόσο δύσκολο ήταν και πόσο θετική ήταν η αντίδρασή σας για το ερώτημα που θέσατε για τις υφιστάμενες ε, διμερείς επενδυτικές ε, συνδίκες που υπήρχαν και πριν ε, από την ένταξη κάποιων χωρών στην Ένωση είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. και αποφασίσαμε να το αγνοήσουμε αυτό το ζήτημα, το βάλαμε κατά το χαλί και τώρα το αγνοούμε για δεύτερη φορά. Νομίζω πως δεν ε, μπορούμε να συνεχίσουμε να αγνοούμε αυτό το ζήτημα γιατί είναι ασύμβατο με την ιδέα μιας ε, κοινή αγοράς να έχουμε διαφορετική μεταχείριση των ε, κρατών μελών της Ένωσης όσον αφορά την προστασία των επενδύσεων. Δεν μπορεί να τα γνωρίσει πλέον το Κοινοβούλιο και σας ευχαριστώ που το θέσατε πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Είναι κάπως περίεργο να αγνοούμε σκεμμένα κάτι το οποίο είναι κλειδί όσον αφορά την ιδέα της ε, εσωτερικής αγοράς. Ας περάσουμε στην ε, ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε από την τροπολογία αριθμός 1. 1 και 16 που είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 54 άρχεται η ψηφοφορία κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται Τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Αντιρρήσεις. Ε, ωραία. Το ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε προφορικά. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 καταπίπτει 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ καταπίπτει. Συγγνώμη. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Ψηφοφορία σε τμήματα. Τμήμα 1. Τη 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 τη 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Α, 99. Να ελέγξουμε την 99. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Ποιος ζήτησε τον έλεγχο. Ο συντάκτης τροπολογίας φυσικά. Οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 102 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Εκατόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν έντεκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν δώδεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 116 ηλεκτρονικά υπέρ. Ε, συγγνώμη, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν έχει ναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 118. Συγγνώμη, 119 υπέρ. Κατά αποχέση απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ 20, συγγνώμη, 20. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 η... σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε την 29 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 29 ναι άρχεται η ψηφοφορία Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. οι συνήθεις μεσολαβητές 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ, σε δύο τμήματα, συγγνώμη. Υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Όχι, τμήμα 1 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τμήμα 1 έρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τμήμα 2 υπέρ τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 κατά πίπτη 35 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αυτό εδώ αντιβαίνει τα πολιτικά μαθηματικά αυτού του κοινοβουλίου. 32. Καταπίπτει επίση. Όχι, όχι. Δύο. Α, η, η δύο, η τροπολογία δύο του εισηγητή. Υπέρ. Τροπολογία δύο. Τροπολογία δύο. Ας επαναλάβουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τριάντα επτά εγκρίνεται. Τριάντα οκτώ, τριάντα εννιά καταπίπτουν. Σαράντα λοιπόν. Σαράντα. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά 42 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τώρα έμαθα. 44 υπέρ, 45 ε, συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και εδώ Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία των τροπολογιών, τελική ψηφοφορία για την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 3, συγγνώμη, 24 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές. Ας ψηφίσουμε για το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, 24 υπέρ, 3 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια στον Παύλ Ζαλεύσκη, στον οποίο θα δώσω τώρα το λόγο, διότι μου το ζήτησε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι που υποστηρίξατε αυτό το φάκελο. Η προτάση μου είναι να πάμε στην Ολομέλεια και να ψηφίσουμε τις τροπολογίες και μετά να ξεκινήσουμε το τριμερή διάλογο πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία πρώτης ανάγνωσης στην Ολομέλεια. Καλώς. Πρέπει να το ψηφίσουμε για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις πριν ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση. Η έγκριση θα είναι η εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Θα συμμετέχει ο πρόεδρος, ο συγητής, η Σκιώδης, David Μάρτιν, από τους σοσιαλιστές, Ιωάννα Βάρνα από την Άλντε, Ζεραντήλ από το ECR, Φρανσίσκα Κακέλερα από τους Πράσινους, Σόλτς από την ΚΟΕ, και κάποιος ακόμα που θα μας πει FD. Ε, Λάγκε, αντερήσεις. Κύριε Πρόεδρε, εγώ είχα καταλάβει αλλιώς την πρόταση του εισηγητή ότι θα πάμε με την έκθεση στην Ολομέλεια, θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες στην Ολομέλεια και μετά θα πάμε στην διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο και τελική ψηφοφορία δεν θα γίνει στην Ολομέλεια, αλλά θα διαπραγματευτούμε. Αλλά θα φέρουμε τις τροπολογίες στην Ολομέλεια. Correct. Mm-hmm. Σωστά. Ναι, σωστά. Εγώ έκανα λάθος. Όντως, ολομέλειες και όχι το τελικό ψήφισμα. Η εντολή, λοιπόν, θα είναι η ψηφοφορία που θα κάνουμε στην Ολομέλεια. Σωστό. Μια στιγμή, Πρόεδρε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αλλά εγώ έχω μείνει λίγο πίσω. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς προτείνεται. Προτείνουμε τη συνήθη διαδικασία για να ολοκληρωθεί η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Έχουμε τις τροπολογίες, θα ξαναψηφιστούν στην Ολομέλεια. Δεν θα ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση, γιατί προτείνει ο συνάδελφος και εφόσον το εγκρίνει και η Επιτροπή μας, να μην έχουμε τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Οπότε Αναβάλλεται η ψηφοφορία στην Ολομέλεια και αρχίζουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με εντολή από τις τροπολογίες που θα ψηφίσει η Ολομέλεια. Έτσι θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν της πρότασης αυτής, αυτού του διακανονισμού. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ, ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. 28 υπέρ, 2 ψήφοι κατά και μία αποχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. floor our voting time has not yet... Δεν έχει λήξει η ψηφοφορία ακόμα, αγαπητοί συνάδελφοι, σημείο 22 τώρα στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για γνωμοδότηση. Για παρακολουθήστε με λίγο παρακαλώ. Είναι γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Μεταφορών. Ο εισηγητής μας είναι ο Ρόμπερτ Στέρντι και πρόκειται για την εξωτερική πολιτική για την αεροπορία της Ευρωπαϊκής Άνωσης. Υπάρχουν 16 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην έκθεση αυτή, στην γνωμοδότηση αυτή, αλλά υπάρχουν και συμβιβαστικές που έχει συμφωνήσει ο εισηγητής με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ο Ρόμπερτ Στέρμπι θα μας τα εξηγήσει. Δεν πρόκειται απλώς ε, μόνο για τι συμβαστικέ τροπολογίε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω του σκιώδει εισηγητέ. Έχω πολλά χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συχνά δυσκολεύομαι στη συνεργασία. Αυτή τη φορά, και συνήθω συμβαίνει αυτό στην Επιτροπή μα, μπορέσαμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά και να καταλήξουμε σε κάτι που πιστεύω εγώ ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ακόμα και Γιάννη και εκεί χαμογελάει δεν συνηθίζει. Ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξή σας. Οι μεταφορές έτσι θα μπορέσουν να λάβουν υπόψη τους τις δικές μας θέσεις. Άλλες φορές δεν συμβαίνει, αλλά αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα βοηθήσει και ότι θα λάβουν υπόψη τους τις δικές μας θέσεις. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ όλους, Πρόεδρε. Πρόεδρος, καλώς. Είναι καλό να ακούμε τέτοια θετικά σχόλια για την συνεργασία μας προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς. Αρχίζουμε την ψηφοφορία λοιπόν τώρα. Τροπολογία 1, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε την τροπολογία 2. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη υποφορίας. Απορρίφθηκε. 22 κατά. 9 υπέρ. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, Δεν ε, ήμουν αφηρημένο. Ξανά παρακαλώ. Ή μάλλον θα ελέγξουμε για την τροπολογία 11. Ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές θα ε, πρέπει να έχει περάσει, αλλά ε, να ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 16. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Έκλεισε. Πέραν η ψηφοφορία και απορρίφθηκε. Οι πολιτικές ομάδες πρέπει να προσέξουν περισσότερο την αριθμητική τους. Δεν είναι λογικό βάσει τη σύνθεση της Επιτροπής αυτή τέλο πάντων. Τελική ψηφοφορία τώρα. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη γνωμοδότηση ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Μπλε, γιατί μπλε, λέει ο πρόεδρος. Πέρα στις ψηφοφορίες. Τώρα. 26 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον Ρόμπερτ Στέρμπι. Και έτσι έληξε η ψηφοφορία. Excellent. My people tell me that you were excellent. They were, they were excellent. Thanks.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 Please, colleagues, this is... Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ε, τελείωσε και η συνεδρίασή μας γιατί έχουμε ένα ανεξέχοντα προσκεκλημένο που θα ακούσουμε σήμερα. Γι' αυτό μη φεύγετε από την αίθουσα παρακαλώ. Οι όλοι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, παρακαλώ, φροντίστε. Let's to item... Περνάμε στο επόμενο σημείο. Λοιπόν, για παρακαλώ, εδώ, καθίστε και προσέξτε με. Επιτρέψτε μου εδώ να καλωσορίσω τον κύριο Ρενό Σοριέλ, ο οποίος είναι γραμματέας της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, ο οποίος δέχτηκε να έρθει εδώ από τη Βιέννη για να μας παρουσιάσει την Επιτροπή αυτή των Ηνωμένων Εθνών, που ασχολείται με την προετοιμασία και την προώθηση του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου. Εμείς είμαστε Επιτροπή Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεπώς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει να μας πει, διότι το εμπόριο είναι μια δραστηριότητα που βασίζεται σε κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μας με τους εταίρους μας ανά τον κόσμο. Σίγουρα θα λάβουμε υπόψη μας τόσα θα μας πει πριν αποφασίσουμε διάφορα θέματα, είτε πρόκειται για την επίλυση διαφορών, είτε πρόκειται για τη διαφάνεια, είτε πρόκειται για τη διατησία βάση συνθήκων ή άλλα νομικά ζητήματα που μας απασχολούν, ε, είτε πρόκειται για την ηλεκτρονική διαβίβαση αρχείων, είτε για διασυνοριακές ε, εμπορικές συναλλαγές κλπ. κλπ. Έχουμε κάθε συμφέρον λοιπόν να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με την Επιτροπή αυτή των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη φορά πάντως που τον έχουμε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που βρίσκεστε εδώ και έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τα μέλη της Επιτροπής αυτής που έχουν το κουράγιο να μείνουν εδώ για να ακούσουν ε, μια γενική παρουσίαση για την Επιτροπή μας των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπόριο. Με την άδειά σας, Πρόεδρε, και με την άδεια των διερμηνέων θα παρουσιάσω στα αγγλικά. Μην ξεχνάμε Βέβαια ότι από την άλλη είμαστε στην επομένη της ημέρας για την ε, γαλλική γλώσσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα αγγλικά είναι η κύρια γλώσσα του οργανισμού που εκπροσωπώ. Ναι, ναι, αλλά τα γαλλικά είναι μια γλώσσα εργασίας εδώ. Ναι, λέει ο κύριο Σοριέλ, είναι μια γλώσσα εργασία, αλλά δυστυχώ διαπιστώνουμε ότι η δουλειά μα κατά το 95% γίνεται στα αγγλικά, 3% στα ισπανικά, 1% στα γαλλικά και τα υπόλοιπα είναι ρωσικά, αραβικά και κινέζικα. Εάν ε, μου επιτρέπετε τώρα να μιλήσω αγγλικά, σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας ε, λόγια. Είναι για εμάς τιμή να είμαστε εδώ πέρα σήμερα και να μιλήσουμε για την πολύ σημαντική επιτροπή του ΟΗΕ, την οποία εκπροσωπώ, τη Διεθνή Επιτροπή για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Ε, σας είμαστε ευγνώμονες για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη δουλειά μας και βεβαίω αναμένουμε να ε, οικοδομήσουμε περαιτέρω την συνεργασία που είχαμε τα τελευταία χρόνια στο θέμα του διεθνούς εμπορικού δικαίου. Βεβαίω να πω πως η σχέση εργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θα μπορούσε να είναι καλύτερη και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Υποθέτω πως λίγα ξέρετε στην αίθουσα για το την καθημερινή πρακτική της Επιτροπής μας και το τι κάνει. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν θα ξεκινήσω με μια γρήγορη παρουσίαση ε, για το ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Η Ανσίτραλη είναι μια γενική, ένα φορέας της Γενικής Συνέλευσης ε, στο σύστημα του ΟΗΕ, δημιουργήθηκε το 1966 με στόχο να συνεισφέρει στην εναρμονισμό και εξυγχρονισμό του, διεθνού, του δικαίου, του Διεθνού εμπορίου. Και βεβαίω ε, πολύ γρήγορα ε, ετέθη το ζήτημα του εξυγχρονισμού του Διεθνού εμπορικού δικαίου. Έτσι τώρα είναι ο βασικός φορέας ε, του ΟΗΕ στο πεδίο του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου με μια γραμματεία στη Βιέννη. Ε, είμαστε μικρός οργανισμός και σχετίζεται με το Γραφείο Νομικών Υποθέσεων του ΟΗΕ και εγώ έχω την τιμή να είμαι διευθυντής ε, της διεύθυνσης του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και της Γραμματείας. Έχουμε εμπειρία 45 ετών στην διαπραγμάτευση και σύνταξη κειμένων, δηλαδή συμβάσεις, υποδείγματα νομοθεσίας, νομοθετικούς οδηγούς σε πάρα πολλούς τομείς. Έχουμε αυτή τη στιγμή έξι διακυβερνητικές ε, ομάδες εργασίας με αντικείμενο την διαπραγμάτευση κειμένων σε εξής τομείς. Δημόσιες προμήθειες, διεθνή εμπορική διαιτησία, επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό εμπόριο, διασυνοριακή χρεοκοπία και ε, ασφαλείς ε, συναλλαγές. Πέρα από αυτά τα έξι θέματα που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, η Ανσίτραλ επίσης ε, έρευνα διάφορα πράγματα. Είχαμε πρόσφατα ένα συμπόσιο για το ζήτημα της μικροχρηματοδότησης ή όπως το λέει ο ΙΕ, ε, το θέμα της, ε, συμπερι, της οικονομικής συμπερίληψης. Και θα έχουμε βεβαίως ε, και μια σχετική πρωτοβουλία που θα αφορά απλοποιημένες μορφές εταιρεία, ε, ειδικά στην Λατινική Αμερική. Επίσης, η Ανσιτράλ ε, είναι ο θεματοφύλακας πολλών συνθήκων στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. πιο, τα πιο γνωστά μέσα είναι η Σύμβαση του 1958 της Νέας Υόρκης για την ε, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων που είναι η θεμέλια λήθος της ε, διαιτησίας όπως λειτουργεί σήμερα. Το άλλο σημαντικό κείμενο που δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε είναι η Σύμβαση του 1980 της Βιέννης για την Διεθνή Πώληση Αγαθών. Και θα επανέλθω σε αυτό όταν θα μιλήσουμε για τη μελλοντική μας εργασία στον τομέα αυτών. Με τα θέματα αυτά και θα επανέλθουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα με την ιστορία και την πρακτική της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να επιμείνω στη διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ του έργου του δικού μας και του έργου του ΠΟΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η δική μας η εντολή είναι αρκετά διαφορετική από αυτή του ΠΟΕ, υπό την έννοια πως ε, εμείς ε, δεν ανησυχούμε τόσο με το να θεσπίζουμε εμπορικούς κανόνες ε, που ισχύουν μεταξύ κρατών δεν θα δείτε ποτέ συζήτηση σε εμάς για τους ε, δασμολογικούς φραγμούς. Επίσης, αντιλαμβάνεστε πως η Ancestral δεν είναι φορέας επίλυσης διαφορών. Ε, ε, δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της νομοθεσίας, αλλά από μόνο μας δεν επιλύουμε διαφορές α, όπως ο καμιά φορά είναι δύσκολο να αντιληφθούμε την ε, αλληλεπικάλυψη αφενός ε, ζητημάτων που αφορούν και την Επιτροπή μας και τον ΠΟΕ παραδείγματος χάρη οι προμήθειες και την θεμελιώδη διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ των δύο οργανισμών. Ως, για όσους είναι οικονομολόγοι, νομίζω ως ένα βαθμό θα σας βοηθήσει να σκεφτείτε την διάκριση μεταξύ μακροοικονομίας και μικροοικονομίας. Δηλαδή ο ΠΟΕ ασχολείται με την ευρύτερη, για τη γενική εικόνα και τις διακρατικές σχέσεις. Η Ancestral προσεγγίζει τα πράγματα όχι από τη σκοπιά α, του, ε, της μίας ρυθμιστικής αρχής που απευθύνεται σε άλλες ρυθμιστικές αρχές. Εμείς προσεγγίζουμε το διεθνές εμπόριο από τη σκοπιά της μικροοικονομίας θα έλεγα, της μεμονωμένης εταιρεία η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες οι οποίες προκύπτουν από τις διαφορές ε, στους νόμους του διεθνούς εμπορίου όταν προσπαθούν να βγουν στις διεθνείς αγορές. Οπότε αυτό έχει σημασία για να αντιληφθούμε τη ρεαλιστική προσέγγιση που έχουμε εμείς, ε, δηλαδή ε, δεν έχουμε θεωρητικά σύνορα όπως στις χώρες στις οποίες παραδείγματος χάρη ε, εντός των χωρών υπάρχει αυστηρή διάκριση μεταξύ αστικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και τα λοιπά. Μπορούμε να ασχοληθούμε με τις δημόσιες προμήθειες, οι οποίες σε πολλές χώρες θεωρούνται περίπτωση του δημοσίου δικαίου λόγω της σημασίας που παίζουν οι δημόσιες προμήθειες, παραδείγματος χάρη, στην καθημερινή διεξαγωγή του εμπορίου από τη σκοπιά της κάθε μεμονωμένης εταιρεία, κάτι το οποίο δεν σημαίνει πως τα αποτελέσματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά του ΠΟΕ. Αλλά είναι διαφορετική η οπτική γωνία όπως σας είπα και είναι σαφές πως τα υποδείγματα νομοθεσίας που έχουμε υπάρχουν πράγματι ε, ουσιαστικές διαφορές μεταξύ του τι κάνει ο ΠΟΕ και της προσέγγισης της δικής μας. Τώρα, πρέπει να ξεκαθαρίσω πως ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του οργανισμού μας η μόνη δραστηριότητα του οποίου είναι να συντάσει νομοθεσία, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά μας είναι πως κανένα από τα προϊόντα μας δεν είναι δεσμευτικό. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε όταν εξηγούμε την Ancestral σε τρίτους ή στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Δεν έχουμε το πλεονέκτημα να βασιζόμαστε σε, μέση, σε μέσα τα οποία γνωρίζουν οι περιφερειακοί οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο Οργανισμός για την Εναρμόνιση του Εμπορικού Δικαίου της Αφρικής. Και οι δύο αυτοί οργανισμοί μπορούν να συντάξουν οδηγίες, κανονισμούς ε, ή ενιαίους νόμους όπως λέγονται, οι οποίοι ε, έτσι ισχύουν στην ένωμη τάξη των κρατών μελών. Στην περίπτωσή μας, επειδή είμαστε οργανισμός του ΟΗΕ, δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός για να φροντίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του προϊόντος της εργασίας μας. Είναι μια δυναμία αυτή την οποία έχουμε προσπαθήσει να μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα και αν δείτε τον οργανισμό μας μετά από 45 χρόνια δραστηριότητας, ε, ο μόνος λόγος για τον οποίο ανησυχεί κανείς για το τι κάνουμε εμείς κάποιοι δικηγόροι σε μια γωνίτσα εκεί του ΟΗΕ είναι το ότι κάποια από τα προϊόντά μας εφαρμόζονται και είναι σε θέση να επηρεάσουν το νομικό πλαίσιο των ε, εμπορικών συναλλαγών. Παγκοσμίω ανέφερα πριν τα παραδείγματα τη σύμβαση τη Νέα για τη Διαιτησία. Είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα πραγματικά ενός ε, παγκοσμίου κειμένου. Πλησιάζουμε τα 215 κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο σημαίνει πως με την εξαίρεση κάποιων χωρών όπως της Μιανμάρ η οποία προσεχώς θα κυρώσει και αυτή τη συνθήκη. Ε, ουσιαστικά όλες οι χώρες με ουσιαστικό και σημαντικό εμπόριο είναι ε, μέλη της συνθήκης. Επίσης, ε, να αναφερθώ στην Σύμβαση του 1980 της Βιέννης για τις πωλήσει με τις πρόσφατες κυρώσεις της Ιαπωνίας πριν από λίγα χρόνια και της Βραζιλίας ε, φέτος, νομίζω πως λίγες χώρες πλέον ε, δεν έχουν ε, υπογράψει. Και με την σημαντική εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ινδίας, όλες οι μεγάλες εμπορικές χώρες είναι μέλη της Σύμβασης του ΟΗΕ για τις πωλήσει και άρα υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί 75 έως 80% του παγκοσμίου εμπορίου. Είπα πως ε, τα προϊόντα μας σε γενικές γραμμές λειτουργούν ε, στην πράξη. Πρέπει επίσης να επιμείνω στο ότι είναι μάλλον επιτυχή γιατί η Ancestral είναι η μοναδική πηγή ε, ενό δικαίου παγκοσμίου στο βαθμό που δέχεται παγκοσμίου δικαίου στο βαθμό που δέχεται κανείς πως κάτι, γίνεται, κάτι μπορεί να γίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων περιφερειακών οργανισμών, δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί φορείς που να παράγουν παγκόσμιο δίκαιο και η Ανσιτράλ είναι ένας από αυτούς. Με επιτυχία όχι μόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπως φαντάζεστε μέρος των λειτουργιών μας είναι το να δίνουμε στον ανθρώπινο κόσμο εργαλεία που δίνουν σε νέες χώρες, χώρες σε μετάβαση, χώρες που για διάφορους ε, λόγους αναζητούν τρόπους εξυγχρονισμού της εμπορικής τους νομοθεσίας. Ε, τους δίνουμε λοιπόν κάποιες προδιαγραφές ε, που βασίζονται σε μια συνένεση και γενικά θεωρούνται ποιοτική νομοθεσία και γενικώς απολαμβάνουν υποστήριξη σε κάθε γωνιά του κόσμου, αλλά δεν κάνουμε μόνο αυτά. Εάν δείτε το τι γίνεται π.χ. στην ε, εμπορική διαιτησία, είναι σημαντικό το ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το να υιοθετούν τις δικές μας προδιαγραφές ε, και αναθεωρούν την ομοθεσία τους με βάση αυτά τα οποία λέμε και με το να εφαρμόζουν τις προδιαγραφές αυτές όχι μόνο για τις διεθνείς συναλλαγές αλλά και για τις εσωτερικές στην περίπτωση της διετησίας με τους πρόσφατους νόμους της Ισπανίας και της Ιταλίας ε, νομίζω πως ε, αναδεικνύεται εδώ πέρα μία τάση λίγα λόγια για την σύνθεση της Ανσετράλ αυτή τη στιγμή έχουμε 60 κράτη-μέλη που έχουν επιλεγεί μεταξύ των κρατών μελών της Γενικής Συνέλευσης με ε, σκοπό να υπάρχει μια ίση εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών ομάδων, όλων των σταδίων της ανάπτυξης, όλων των ειδών τα νομικά συστήματα και γενικώ ε, όλες τις συνθήκες μπορούν να βρεθούν διεθνώς. Ενδιαφέρον ναι, για εσάς ε, είναι το ότι υπάρχουν 14 κράτη-μέλη από την ομάδα Δυτικής Ευρώπης και λοιπόν και 8 χώρες από την ομάδα Ανατολικής Ευρώπης και, Ανατολικής Ευρώπης και λοιπόν. Υπάρχουν δηλαδή 10 με 12 κράτη-μέλη ανα πάσα στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στον Ανσιτράλ ε, ως μέλη της Ανσιτράλ ε, είτε ως μέλη της ε, ομάδας Δυτικής Ευρώπης είτε ως μέλη της ομάδας Ανατολικής Ευρώπης. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην σχέση μεταξύ της Ανσιτράλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπα, υπάρχει περιθώριο βελτιώση, αλλά υπάρχει και μια αρκετά εδρεωμένη συνεργασία. Θα θα καλέσω να κοιτάξετε και τις γραπτές σημειώσεις που μοίρασα για πώ πώς θα μπορέσουμε να συνοψίσουμε τα έργα που καλύπτουν οι ομάδες εργασίας μας. Στα λίγα λεπτά που μου απομένουν θα εστιάσω σε λίγα, σε ένα-δύο παραδείγματα το παράδειγμα καταστάσεων συνεργασίας είναι θετικό. Αλλά όταν μιλάμε για δημόσιες προμήθειες, γνωρίζουμε τις προσπάθειες ε, που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι τεχνικές όπως συμφωνίες πλαίσιο ηλεκτρονικές ε, αντίστροφοι, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, ε, δηλαδή χαρακτηριστικές ε, ευρωπαϊκές οδηγίες, έχουν υιοθετηθεί με κάποια τροποποίηση από το Αντιστρόλ και από χώρε άρα πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια από αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται και από τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες στον τομέα δημοσίων προμηθειών υψηλής αξίας ε, υποδομών. Βρίσκουμε εκεί πέρα διαφορετικά στοιχεία του ε, διαλόγου του ανταγωνιστικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εναρμόνιση των διαδικασιών λοιπόν δεν ενισχύει μόνο την διασυνοριακή εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων αλλά προωθεί και ε, την διάδοση προδιαγραφών. Από το 2004 έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι διαφορές των προδιαγραφών Ανσετραλ και Ευρωπαϊκής Ένωση Άρα χώρε οι οποίες αναζητούν οικονομική στήριξη ή ανάπτυξη υποδομών είτε από τις ε, τράπεζες ανάπτυξης είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνουν με βάση παρόμοιε προδιαγραφέ. Αν δούμε τώρα τα τη χρεοκοπία. Ε, σας παρακαλώ πάλι να ρίξετε μια ματιά σημειώσεις μου. Αλλά σημαντικό είναι να ξέρουμε πως υπάρχει μια σχέση μεταξύ των ζητημάτων αυτών που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και των όσων κάνουμε εμείς στο παγκόσμιο επίπεδο. Η σημασία της ε, νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ερμηνεία του υποδείγματος νομοθεσίας μας ε, ορίζεται και φαίνεται και σε εγχειρίδιο που έχουμε εκδώσει και είναι ένας οδηγός εφαρμογής. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω για την σημασία που έχει η ε, ενιαία ερμηνεία το, της υποδειγματικής αυτής νομοθεσίας. Αν δείτε τώρα τα της διαιτησίας, να σας πω πως γενικά η συνεργασία είναι καλή έχουμε υψηλό επίπεδο συμμετοχής ε, των ε, ευρωπαϊκών χωρών ε, στην αναθεώρηση του υποδείγματος νομοθεσίας για την διαιτησία. Πέρα από εκεί έχουμε καλή συνεργασία στον τομέα της εμπορικής διαιτησίας. Η οδηγία που υιοθετήθηκε το 2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γενικές γραμμές ε, συμφωνεί και είναι σύμβατη με το δικό μας υπόδειγμα νομοθεσίας και το ε, πιο πιο η συνεργασία είναι σε ένα τομέα που δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει συνεργασία μας και θα σας ενδιαφέρει είναι ο τομέας της διαφάνειας στην διαιτησία σε περιπτώσει όπου υπάρχει κάποια ε, σύμβαση, σε περιπτώσει επενδύσεων. Οι εκπρόσωποι σα εμπλέκονται ενεργά στην ομάδα εργασίας παριθμών 2 για νομικές προδιαγραφές για τη διαφάνεια και το κείμενο αυτό όπως μάλλον ξέρετε μόλις εγκρίθηκε ε, στην Νέα Υόρκη από την ομάδα εργασία και αναμένουμε να οριστικοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι φέτος. Η οδηγία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2012 επίσης αντικατοπτρίζει ένα σημαντικό κανονισμό για τις διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες και προσφέρει νομική ασφάλεια σε διμερείς ε, συμφωνίες επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Αναμένουμε οι επενδυτικές συμφωνίες της Ένωσης να κάνουν λόγο ε, για τους κανόνες αυτούς όσον αφορά την διαφάνεια στην επίλυση διαφορών. Επίσης, να επισημάνω πως υπάρχει μια πρόταση της Ανσιτράλ για τη σύσταση ενός μητρώου για την στήριξη της ε, λειτουργίας των κανόνων διαφάνειας και έχουμε κάποιες συζητήσεις για να αξιολογήσουμε το πιθανό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη στήριξη αυτού του Μητρώου. Αν δούμε τώρα κάποιους τομείς όπου υπάρχουν, υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης συνεργασίας. Θα πω λίγα γρήγορα πράγματα για το ηλεκτρονικό εμπόριο Πρόκειται για ένα τομέα όπου έχουμε ενεργή συνεργασία τα τελευταία 20 χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ανσιτράλ ήταν ε, πρωτοπόροι στον τομέα αυτών. Θα έλεγα δε πως ε, εδώ πέρα αποδεικνύεται η δυσκολία και των δύο οργανισμών στο να καταλήξουν σε μία μέθοδο εργασίας ε, που θα επιτρέπει την ε, ειλικρινή ανταλλαγή πληροφοριών. Γιατί εμείς επηρεαζόμασταν από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο ναι, αλλά και αντιστρόφως βεβαίω. Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια σχέση εργασίας για ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών μεταξύ κομισιών αφενός και της γραμματείας μας αφετέρου ε, κάτι το οποίο νομίζω θα αφελούσε και τους δύο οργανισμούς μας. Αυτή τη στιγμή ε, ένα σημείο που μας δυσκολεύει ακόμα είναι το θέμα της σύμβασης ε, του ΟΗΕ του 2005 για την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου στο διεθνές εμπόριο. Το κείμενο αυτό δεν έχει βρει ακόμα στήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρά το ότι περιέχει μια ρήτρα από σύνδεσης που στόχο έχει να διατηρήσει την αυτονομία του ευρωπαϊκού δικαίου. Και βεβαίως θα πρέπει να κρίνουμε άπαξ και διαπαντός το εάν επαρκεί αυτή η ρήτρα ή το τι άλλο μπορούν να κάνουν από κοινού οι δύο οργανισμοί μας έτσι ώστε το κείμενο αυτό να στηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όπως θα έπρεπε. Τέλος θα αναφερθώ στο ε, δίκαιο των συμβάσεων. Το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τελευταία επικαλύπτεται με το δικό μας. Το τελευταίο έτος η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων εξέτασαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πολίσεων. Μάλιστα, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έκανε και μια δημόσια ακρόαση την τρίτη που μας πέρασε πριν δύο μέρες για το θέμα αυτό. Η πρόταση αυτή που δεν έχει εξεταστεί από ό,τι καταλαβαίνω από την Επιτροπή σας ακόμα πρότεινε ένα εναρμονισμένο περιφερειακό καθεστώς συμβάσεων για διοσυνοριακό εμπόριο ε, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Επικεντρώνεται σε συναλλαγές λιανικής και μικρομεσαίε επιχειρήσεις, παρά το ότι το πεδίο εφαρμογή αυτή τη στιγμή είναι ακόμα ανοιχτό. Το σκεπτικό λοιπόν της πρότασης αυτής ε, είναι ε, το γνωστό, ότι δηλαδή οι διαφορές στην ομοθεσία μεταξύ των χωρών μπορούν να αποθαρρύνουν τους εμπόρους και τους καταναλωτές από το να κάνουν ε, διασυνοριακές διαλέγες. Αν υπάρχει λοιπόν ένα ενιαίο δίκαιο δεν θα υπάρχει αυτή αυτή, αυτός ο αποτρεπτικός παράγοντας, ούτε ε, το επιπλέον κόστος. Η πρόταση της Κομισιόν ενδιαφέρει την Ανστραλ και φαντάζομαι και την Επιτροπή σας, γιατί αφορά το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, ειδικά την αποτελεσματικότητα της διεθνούς εναρμόνισης και μηχανισμών όπως η Σύμβαση για τις πωλήσει του ΟΗΕ και παρά το ότι η Άνσιτραλ δεν είχε εμπλακεί στην ανάπτυξη της πρότασης της ε, Κομισιόν. Πάρα πολλές από τις ε, διατάξεις ε, της πρότασης εμπνέονται από την Σύμβαση Πολίσεων της Βιέννης. Οι βασικές διαφορές είναι πως η Σύμβαση Πολίσεων είναι ένα διεθνές μέσο και περιορίζεται σε εμπορικές και όχι λιανικές συναλλαγές και συγκεκριμένα αφορά την πώληση αγαθών. Η σύμβαση λοιπόν της Βιέννης για τις πωλήσει ε, έχει θετηθεί από 79 χώρες και θα μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 9 από τους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους της είναι συμβαλόμενα μέρη μεταξύ των οποίων ΗΠΑ, Κίνα, ε, Ρωσία, Ελβετία και Νορβηγία. Επιπλέον, Συνολικά τα συμβαλόμενα μέρη καλύπτουν το 75% του ε, εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης. Εσωτερικά λοιπόν η συνθήκη αυτή είναι ήδη ε, ε, εσωτερικό, δίκαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 23 από τα 27 κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη εξετάζεται η σύμβαση αυτή για τους λόγους αυτούς. Η συνθήκη για τις ε, συμβάσεις για το διεθνές εμπόριο είναι σημαντικό εργαλείο για τους Ευρωπαίους ε, εμπορευόμενους. Και βεβαίως ε, η σκέψη για την εφαρμογή της και σε πωλήσει πέραν είναι κάτι το πολύ σημαντικό μπορεί έτσι να προωθηθεί το εμπόριο και η ανάπτυξη και να προχωρήσουμε σε περαιτέρω εναρμόνιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο βαθμό όμως που αφορά τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές ε, υπάρχει ο κίνδυνος να περιπλακεί η, η διεπιστάμενη Το σημειώσαμε αυτό με ανησυχία πέρσι στην δική μας την σύνοδο πως το να προσθεθεί άλλο ένα περιφερειακό επίπεδο στο διεθνές καθεστώς πώλησης αγαθών θα μπορούσε να διαταράξει την εναρμόνιση που έχει ήδη επιτευχθεί. Όπως έχει αυτή τη στιγμή η πρόταση μπορούμε να φανταστούμε έναν Ευρωπαίο έμπορο ο οποίος θα αντιμετωπίζει τη δύσκολη ε, δυνατό, την δύσκολη, να βρεθεί στη δύσκολη κατάσταση να αντιμετωπίζει τρία διαφορετικά καθεστώτα. Τη σύμβαση αυτή της Βιέννης, ε, το μέσο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Εθνικό Δίκαιο για οποιοδήποτε ζήτημα δεν καλύπτεται από τα δύο προηγούμενα. Το επιπρόσθετο αυτό στρώμα θα σημάνει ένα επιπλέον νομικό κόστος και θα αποθαρρύνει οπωσδήποτε κάποιους. Καθώς εστιάζουμε κυρίως βεβαίως σε συναλλαγές λιανικής και ανάλογες με αυτές, θα πρέπει να μπορεί η γραμματεία μας και τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα να συνεργαστούν έτσι ώστε τα δύο αυτά μέσα να λειτουργούν παράλληλα για να προωθηθεί ένα εναρμονισμένο περιβάλλον για τις πωλήσει στην Ευρώπη και διεθνώς. Αυτή τη στιγμή δεν είχαμε καμία ευκαιρία εμείς να συνεισφέρουμε στη διαδικασία αυτή ελπίζουμε η Επιτροπή σας με την εμπειρία που έχει στο Διεθνές Εμπόριο θα συμπεριληφθεί περαιτέρω κοινοβουλευτικές συζητήσεις ε, που θα αφορούν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζουμε και η Άντσετρα να έχει περαιτέρω ευκαιρίες να συζητήσει το θέμα αυτό που αφορά και τους δυο μας. Τώρα, για να καταλήξω το πρόβλημα, να ολοκληρώσω για να ε, κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Όπως βλέπετε η δικιά μας εργασία κάπου τέμνεται με τη δικιά σας. Θέλουμε και οι δύο να εναρμονίσουμε το διεθνές εμπορικό δικαίο, όχι μόνο προ το συμφέρον των κρατών μελών μας, αλλά και προ το συμφέρον των ε, ανθρώπων και τη οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται βεβαίω στην οικονομική βεβαιότητα, στην νομική βεβαιότητα, με στο διεθνές εμπόριο. Ελπίζω να σας έδωσα λοιπόν μια ιδέα για το ότι υπάρχει δίκαιο και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο Κάποιοι στον ΟΗΕ ε, φροντίζουν με έναν τρόπο κεντρικό και όπως σας είπα αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην εργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ελπίζουμε να συνεργαστούμε αν μας δοθεί ευκαιρία και ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι η παρουσίαση αυτή έχει μοιραστεί σε όλους. αυτά που είπατε. Έχουμε ήδη κάποια έντυπα ενημερωτικά και θα μοιράσουμε και την ομιλία σας. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να συζητήσουμε, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίτλ Γιουλ Τι νομίζετε εσείς ότι υπάρχει πρόβλημα με την αναρμόνιση και τις συναλλαγές. Θέλουμε κάποια αντίδραση. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η αναρμόνιση ή όχι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέτουμε σε κίνδυνο την ε, δουλειά αυτή και τη συνεργασία με την Ιουστράλ γιατί ε, μας βοηθάει η συνεργασία. Εξάλλου η συνεργασία αυτή έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, έχει πράγματι ενισχυθεί. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να αντιδράσω στην παρουσίαση του κύριου Σορέλ και ευχαριστώ και που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας ε, θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Πρώτα απ' όλα να σας πω που ε, μπορεί να υπάρξει ακόμα βελτίωση στη συνεργασία μας και μετά να έρθω λιγάκι στα θέματα της διαφάνειας ε, και θέματα Investor State. Όσον αφορά το δίκαιο πολίσεων, ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις Υπάρχει η τρέχουσα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και εμείς στη Γενική Διεύθυνσή μας με την δικαιοσύνη ε, δουλεύουμε εντατικά για να διευκρινιστούν αυτά τα ζητήματα. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη αρχίσει και βοηθάει και βοηθούν και τα Ηνωμένα Έθνη για να βρεθούμε, να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Επίσης τώρα για το θέμα της επίλυσης διαφορών online. Και εδώ έχουμε υιοθετήσει νομοθεσία όσον αφορά την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια η προστασία του καταναλωτή. Έτσι, αυτό είναι κεντρικό για μας όταν εξετάζουμε τέτοια θέματα και φροντίζουμε και η δουλειά της Συνουστράλη να αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό το στόχο, δηλαδή την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και δεν πρόκειται μόνο για διαφορές ε, καταναλωτών με επιχειρήσεις, αλλά και επιχειρήσεων μεταξύ τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή δουλεύει εντατικά για το θέμα της επίλυσης διαφορών online. Δουλεύουμε ε, βάσει συνένεσης. Πιστεύουμε ότι τα θέματα που παραμένουν θα διευκρινιστούν. Τώρα έρχομαι λιγάκι στον τομέα που αναφέρατε κι εσεί σαν το κύριο παράδειγμα καλή συνεργασία μεταξύ μα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε κι εσεί, γιατί είναι ένα τομέα πάνω στον οποίο έχουμε κι εμεί επενδύσει πολύ από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με δικηγόρου από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Και γιατί, γιατί πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό του Investors of State είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό οι διαφορές στον τομέα αυτό να επιλύονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Γιάννη Σιτράλ δουλεύει στην ομάδα εργασίας 2 για την ε, διαφάνεια και τον διακανονισμό τέτοιων ε, διαφορών. Και εμείς ε, το κάνουμε αυτό και υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Υπάρχει η αρμοδιότητα αυτή σε μας και γι' αυτό συνεργαζόμαστε μαζί σας και με τα κράτη-μέλη προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Όπως είπε και ο κύριος Σορέλ στην παρουσίασή του, επετέθηκε συμφωνία στις αρχές της χρονιάς και ενημερώθηκε και η Επιτροπή σας γι' αυτό. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για την ε, επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες διασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα, τα σχετικά με τη διατησία σε αυτό το τομέα, είναι ανοιχτά προς το κοινό και τα διαφερόμενα μέρη μπορούν και εκείνα να συνεισφέρουν στα δικαστήρια. Υπάρχει μια νομοθετική πρόταση που ψηφίσατε εσείς σχετικά μάλιστα σήμερα και είναι πολύ καλό αυτό γιατί προχωράμε ακόμα περισσότερο στη διαφάνεια για τις περιπτώσεις αυτές διακανονισμού. Τον Ιούλιο φέτος θα υιοθετήσει κάτι και η Γιουνστράλ όσον αφορά τους κανόνες διαφάνειας, τους οποίους και εμείς θα τους χρησιμοποιήσουμε βέβαια για την επίλυση διαφορών κάθε φορά που πρόκειται για επενδυτικές συμφωνίες. Ένα σημαντικό θεσμικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι συμμετέχουμε και εμείς στις διαπραγματεύσεις με μία φωνή ως Ευρώπη. Κάτι το οποίο μας κάνει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και νομίζω ότι αυτό βοήθησε να έχουμε τα καλά αποτελέσματα που είχαμε όσον αφορά την διαφάνεια στην επίλυση διαφορών. Είναι ένα καλό παράδειγμα που δείχνει πού μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο και έτσι θα συνεχίσουμε και εμείς τη συνεργασία μας μαζί με την UNCITRAL αλλά και με τη δικιά σας επιτροπή όσον αφορά την επίλυση διαφορών στον τομέα του Investor State. Από εκεί και πέρα, αν έχετε κάποια ερώτηση, προτιμάω να με ρωτήσετε εσείς και να μην προσθέσω εγώ τίποτα άλλο. Πρόεδρο. Καλώς. Θα έχουμε εξάλλου και άλλες ευκαιρίες. Σίγουρα θα ξανάρθετε να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Ερωτήσεις τώρα. Παρακαλώ. David Μάρτιν από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, δεν έχουμε εμεί ε, ακόμα τίποτα σχετικά με το έργο της Unistral, αλλά φαντάζομαι ότι θα το λάβουμε όπου να είναι. Ε, μου άρεσε που μιλήσατε για τις σχέσεις και με τον ΠΟΕ Βρήκα ενδιαφέρουσα και τα σχόλιά σας όσον αφορά το εσωτερικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση διαφορών, για παράδειγμα. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή. Εγώ βλέπω ξεκάθαρα πώς ε, τα πρότυπα νομοθεσίας και γενικότερα το έργο σας πώς μπορεί να βοηθήσει. Αλλά θέλω να ξέρω πέρα από την παραγωγή αυτή των νομοθεσιών και τα λοιπά, μπορείτε να βοηθήσετε τις αναπτυσσόμενες χώρες με κάποιο άλλο τρόπο πέρα από αυτούς τους κανόνες. Αν μια αναπτυσσόμενη χώρα αναπτύσσει τους δικούς της και εκπονεί τους δικούς της ε, κανόνες για το εμπόριο, εσείς μπορείτε να βοηθήσετε ώστε να διασφαλίσετε ότι αυτή θα είναι συμβατή με το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Και όταν κάνει διαπραγματεύσεις μια χώρα με κάποιον εμπορικό εταίρο, είτε την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε κάποιος άλλος, Ακούμε συχνά από τους διαπραγματευτές των χωρών αυτών των αναπτυσσόμενων ότι δεν έχουν την πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να τους βοηθήσετε εσείς ή μπορείτε εσείς, φαντάζομαι δεν κάνετε διαπραγματεύσεις ε, αντί για αυτούς, αλλά μπορείτε να τους ενημερώσετε για τις συνέπειες, για παράδειγμα, που θα έχει μια εμπορική συμφωνία που ετοιμάζουν πώς θα μπορεί να ερμηνευτεί ενδεχομένως ε, το α ή το β σημείο της συμφωνίας αυτής. Μπορείτε να δώσετε γενικές αλλά και ειδικέ πληροφορίες στις χώρες αυτές όταν προχωρούν σε τέτοιες συμφωνίες. Παρακαλώ, από την ΚΟΕ, κύριο Σόλτς τώρα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την ολοκληρωμένη ενημέρωση σε σχέση με την Uncitral ήθελα να αναφερθώ στην εισαγωγή σας ε, σε και να σας κάνω μια ερώτηση. Ένα από τα καθήκοντα ενό τέτοιου διεθνού οργανισμού στον τομέα του διεθνούς εμπορικού δικαίου αρμόδιου για το συντονισμό μεταξύ ΣΥΤΡΑΛ, ΠΟΕ, UNDP, UNCTAD και ούτω καθεξής τεθεί το ερώτημα το για ποιο λόγο έχουμε κολλήσει στον ΠΟΕ. Και δεν χρησιμοποιούμε διμερεί συμβάσει μεταξύ. και στο πλαίσιο των διμερών συμβάσεων. Η ερώτηση είναι, μπορείτε να επηρεάσετε αναπτύσσοντας νομοθεσία να δώσετε στους εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να αναγνωριστούν σε ισότιμο επίπεδο ως αμοιβαίοι εταίροι αναπτύσσοντας στη συνέχεια ε, συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τις ε, συμβάσεις που έχουν συναυθεί. Αυτό πιστεύω θα ήταν πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό καθήκον της ε, Επιτροπής εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαρίο, έχετε ξανά το λόγο. Α, συγγνώμη. Μαρία Τσαρνέζο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είστε ένας διεθνής οργανισμός σημαντικός Εργάζεστε σε θέμα ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε για ποιο λόγο δεν προχωράτε, για ποιο λόγο δεν υπερασπίζεστε μια ιδέα δεσμευτικής ποιότητα στο πλαίσιο υγειονομικών προτύπων, εργασιακών προτύπων, περιβαλλοντικών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου. Και θα ήθελα να μου πείτε εάν μελετάτε αυτό το θέμα και κατά πόσο προσπαθείτε να προχωρήσουν τα πράγματα ειδικότερα στις σχέσεις με τον ΠΟΕ ζητώντας του να συμπεριλάβει στη συμφωνίες υψηλού επίπεδου, σε προγραμματεύσεις υψηλού επίπεδου, ενδεχομένω στι ελάχιστε προδιαγραφέ και να συμπεριλάβει τέτοια θέματα και στο σύνολο των συμφωνιών διεθνού εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χρονικό περιορισμό. Θα σας ζητήσω λοιπόν να είστε πολύ σύντομο στις απαντήσεις σας σε αυτές τις παρατηρήσεις της Κομισιόν ή στις, και στις ερωτήσεις των συναδέλφων αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαζόμουν ώρες για να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε την Κομισιόν. Έκτιμα με την ε, έκφραση καλή βούληση και πράγματι είναι σαφές ότι η αμοιβαία εργασιακή σχέση μας ε, βελτιώνεται. Μας ανησυχεί το τι θα συμβεί με αυτή την ε, ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, το ODR. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι η Κομισιόν εξετάζει το ζήτημα με πολύ, πολύ απλά μόνο όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών και η προστασία των καταναλωτών ε, εξετάζεται μόνο μέσω της διατήρησης, ε, της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των καταναλωτών να προσφύγουν στα τοπικά δικαστήρια. Εμείς ελπίζουμε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση ένα βήμα παραπέρα και να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ώστε να αντιληφθούμε ότι ουσιαστικά εδώ έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση όπου κανένας τοπικός δικαστής δεν μπορεί να επιλύσει ένα τέτοιο ζήτημα όταν υπάρχει μια συναλλαγή καταναλωτή στην Ευρώπη με έναν πολιτή ας πούμε στην Κίνα ή στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσφύγει κάποιος στο τοπικό δικαστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λύση. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Περνώντα τώρα στην πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση της τεχνικής ε, αρρωγής ε, που εμείς ε, εξετάζουμε μεγάλη προσήλωση είναι φυσικά μπορούμε να βοηθήσουμε χώρες στον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας τους ε, κάνοντας αναφορά στα δικά μας πρότυπα. Αυτό μπορεί να γίνει με χαμηλό σχετικά κόστος. Συνίσταται ουσιαστικά στον έλεγχο ενός ε, σχεδίου που συντάσσεται στην ε, λόγω χώρο. Χρειάζεται μια ελάχιστη ευαισθητοποίηση εκ μέρους της εν λόγω χώρας. Τώρα όσον αφορά, όπως συχνά συμβαίνει, την ε, εκτίμηση του τι είναι ο νόμος σε μια συγκεκριμένη χώρα και αν το θέμα αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης ε, ότι υπάρχει ανάγκη εξυγχρονισμού της νομοθεσίας ώστε η χώρα να πλησιάσει στα επίπεδα του διεθνούς εμπορίου αυτό φυσικά ξέπερνάει κατά πολύ τις δυνατότητές μας. Συγγνώμη. Να είστε παρακαλώ πιο σύντομο, γιατί έχω κι άλλο ένα θέμα και απομένει λιγότερο από μισή ώρα. Πόσα λεπτά έχω, ένα, δύο, ένα, δύο. Συγκεκριμένες οδηγίες εκδίδονται, οι οποίες προορίζονται για τη βελτίωση του τεχνικού επίπεδου των διαπραγματευτών σε αυτές τις χώρες, στο πεδίο, ας πούμε, των 20 συμβάσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή συντονισμός ε, ευρύ ζήτημα. Δεν είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε τίποτα. Προσπαθούμε, αλλά με πολύ περιορισμένα μέσα. Το ίδιο ισχύει μάλλον και για την τελευταία ερώτηση όσον αφορά τον ΠΟΕ, τη σχέση με τον ΠΟΕ, πρότυπα BIT, τα υγειονομικά πρότυπα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι σίγουρα ζητήματα που εμείς δεν εξετάζουμε. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο UNCITRAL είναι μια συμμαχία κρατών μελών, αλλά η γραμματεία της Ανσίτραλ ε, είναι περίπου 25 άτομα, εκ των οποίων νομίζω έχουμε 15 νομικούς. Ε? Με τα θέματα λοιπόν που σας περιέγραψα ήδη, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε υψηλό φόρτο εργασίας και απλά δεν υπαρκούν οι πόροι μας για να αντιμετωπίσουμε τα πολύ σημαντικά ζητήματα που αναφέρθηκαν εδώ. Ευχαριστώ. Πράγματι, μάθαμε πολλά καινούργια πράγματα μέσα από αυτή την επαφή μας και μας ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι είχαμε την ευκαιρία να σας έχουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε ξανά. Περνάμε τώρα στο σημείο 24. Έχουμε λιγότερο από μισή ώρα, αλλά οι δερμηνοί μας, μας πολύ και μας ε, έδωσαν 10 επιπλέον λεπτά. Κινηθούμε λοιπόν γρήγορα. Αφορά το σημείο 24, τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων τώρα με εξωτερικού εμπειρογνώμονε ε, για την πρώτη ετήσια έκθεση τη Επιτροπή προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τι δραστηριότητε των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών. Η συγκεκριτή είναι ο κύριο Γιάννη Ξαντό. Έχετε το λόγο αμέσω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο ώστε να αφήσω το μέγιστο δυνατό χρόνο στους προσκεκλημένους μας και θα ήθελα φυσικά να τους ευχαριστήσω ε, από όπου και αν ε, προέρχονται, ε, από την υπηρεσία εξωτερική δράση, στη Γενική Διεύθυνση Μάρκετ. Σε αυτή τη συζήτηση υπάρχουν κάποιε δυσκολίε σε όλα τα θεσμικά όργανα το να καταλήξουμε κατά κάποιο τρόπο στο να λαμβάνουμε υπόψη θέματα τα οποία δεν είναι εμπορικά. Όπως ξέρετε αυτό που αποφασίζουν τα θεσμικά όργανα είναι ότι τα κράτη μέλη όσον αφορά τι δραστηριότητε των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του, ε, κυρίω με του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο κυρίω 21. Αυτό που είδαμε από τις πρώτες εκθέσεις που λάβαμε είναι ότι τα κράτη-μέλη δυσκολεύονται εξαιρετικά. Δεν αμφιβάλλω για τη βούλησή τους, αλλά δυσκολεύονται. Και το ζήτημα σήμερα είναι το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα, διότι πιστεύω ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις εξωτερικές δράσεις και στη συμμόρφωση αυτών με τους στόχους της συνθήκης, ε, κυρίως της συνθήκης Λισαβόνας. Για άλλη μια φορά λοιπόν ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας που έχουν έρθει εδώ και είμαι βέβαιος ότι θα μας ενημερώσουν ε, και ότι ε, τα όσα θα μας πούν θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις σε αυτή την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε ακούγοντας έναν εμπειρογνώμονα από την Κομισιόν, τον κύριο Μπερνιαπάντα, από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Που βρίσκεστε. Δεν μπορώ να σας δώσω πάνω από 10 λεπτά. Ακατέβατα. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι θα είναι αρκετά είναι φοβερή η ευκαιρία που βρισκόμαι μαζί σας σήμερα. Εργαζόμαι στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, όπου προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών εταιρείων σε θέματα περιβάλλοντος και δικαιωμάτων και αυτό αφορά όλους τους τομείς. Δεν ισχύει όμως απαραίτητα στους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά γίνεται μία προσπάθεια η οποία μπορεί να εμπνεύσει τις σχετικές εξελίξεις που σχετίζονται με τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. Αυτό είναι ένα μέτρο, επαναλαμβάνω, που ισχύει για εταιρείες και όχι κράτη-μέλη. Είναι μια προσπάθεια που εμείς πιστεύουμε που πιστεύουμε έχει μεγαλύτερο νόημα για μεγάλες επιχειρήσεις επειδή είναι σαφές ότι η επιπτώση για το περιβάλλον και για την κοινωνία μας ευρέως σχετίζονται άμεσα με το μέγεθος και την πολλοπλοκότητα των εταιριών και κατά πόσο δραστηριοποιούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Ήδη εδώ και δύο χρόνια εργαζόμαστε στην ανάπτυξη μιας οδηγίας ως νομοθετικού μέσου και ελπίζουμε να την παρουσιάσουμε στο εγγύς μέλλον. Ανακοινώθηκε ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2011 στην ανακοίνωση για την ενιαία πράξη αγοράς και τον Νοεμβρίο εκείνης χρονιάς στην ανακοίνωση για το CSR. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια των επιχειρήσεών μας και η αποκάλυψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών. Αντιληφθήκαμε ότι οι ευρωπαϊκές ε, εταιρείε διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για σχετικές πληροφορίε παρότι αυτές οι περιβαλλοντικές και ε, υπάρχουν περιβαλλοντικές και κοινωνικές προφορίες που δεν έχουν ε, επισημανθεί επαρκώς. Μελετάμε το θέμα, διεξήγαμε μια σειρά διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους, με κράτη-μέλη, με επιχειρήσεις και με κυβερνητικές οργανώσεις θα γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε το Φεβρουάριο δύο ψηφίσματα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που ουσιαστικά αφορούν αυτά τα σημεία και που βοηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα σημαντικό σημείο που θα ήθελα να υπενθυμίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ούτως ή άλλως πρώτη όσον αφορά τη διαφάνεια σε περιβαλλοντικέ και κοινωνικές πληροφορίες. Πουθενάλλου στον κόσμο οι επιχειρήσεις δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένε σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα όσο οι ευρωπαϊκές. Αλλά παραμένει το γεγονός ότι λιγότερες από 3.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη από όσες υπάρχουν ε, αναφέρουν τακτικά ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πληροφορίες. Πολύ μικρό κομμάτι από τις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν το 10%. Αυτή ήταν λοιπόν η διαπίστωσή μας ότι αν θέλουμε αυτό να αφορά όλους τους τομείς, ειδικά και τους τομείς που σχετίζονται με οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, όπως τράπεζ, το τραπεζικός τομέας ή ο ασφαλιστικός τομέας, η πρώτη ας πούμε κάθε τομέα σε κάθε κράτος μέλος γνωρίζουν, αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της διαφάνειας σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα αλλά οι μικρότερες εταιρείες ε, δεν έχουν υθετήσει τέτοια προσπάθεια. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη μείωσης του φόρτου και αποφυγή του φόρτου προς τις εταιρείε όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό το λόγο δεν θα έχουμε μια υπερβολικά δεσμευτική προσέγγιση σε αυτό την νομοθεσία. Θα φέρουμε τεράστιο περιθώριο ευελιξία για τις εταιρείε, οι οποίες θα μπορούν να επιλέγουν να υποβάλουν εκθέσει με τον τρόπο που θεωρούν καταλληλότερο πιο καλά προσαρμοσμένο στις δικές τους ανάγκες και να παρουσιάζουν μια εικόνα των δραστηριοτήτων τους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά επίσης πιστεύουμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα διεθνή πρότυπα όπως ε, το Global Compact των ε, Ηνωμένων Εθνών ε, και τα πρότυπα για τις πολυεθνικές εταιρείες. και το GRI που επίσης βοηθά σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες ε, σε εθνικό επίπεδο, όπως το Carbon Project, που βοηθά ιδιαίτερα στον τομέα των εκπομπών άνθρακα, ειδικότερα. Αλλά ουσιαστικά στόχος εδώ δεν είναι να επικυρώσουμε, να εγκρίνουμε οποιοδήποτε από αυτά τα πλαίσια, αλλά να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες να τα λαμβάνουν υπόψη με τον τρόπο που θεωρούν πιο χρήσιμο για αυτές. Για να ολοκληρώσω θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο σαφή μηνύματα. Το πρώτο ότι αυτό το μέτρο αφορά ωφέλιμες, χρήσιμες πληροφορίες για τις εταιρείες αλλά και για τους μετόχους, τους επενδυτές γενικότερα καθώς και για την κοινωνία των πολιτών γενικότερα. Ωφέλιμες, χρήσιμες πληροφορίες ε, ισχύει για εφαρμόζεται σε μεγάλες εταιρείες και ότι δεν θα επιβληθούν νέες απαιτήσει για ε, επιχειρήσεις ευρωπαϊκής κλίμακας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Τόμπια Σκίν. Από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός 1233 του 11 προβλέπει την συμμετοχή της, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης με στόχους την σταθερότητα της δημοκρατικής αξίας κτλ. Αλλά κυρίως να εφαρμόζεται το σύστημα των εξαγωγικών πιστώσεων στις διάφορες εμπορικές δραστηριότητες. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, πάντως βάσει του κανονισμού αυτού, λέει ότι η συνθήκη Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το άρθρο 21 δηλαδή της συνθήκης, μπορεί να χρησιμεύσει ως πλαίσιο για να μπορούμε να εξολογούμε τις πολιτικές ε, και των διαφόρων κρατών μελών όταν προχωρούν σε εξαγωγικές επιστώσεις. Τώρα, τι εργαλείο πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς και τι κριτήρια μπορούμε να αναπτύξουμε. Είναι κάτι το οποίο ήδη κάνει ο ΩΣΑ, ήδη από το 2005, όπου υιοθέτησε μία σύσταση για κοινή προσέγγιση όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις που λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικές, ε, για παράδειγμα, παραμέτρους ή και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων επίσης χρησιμεύει. Τώρα, στην ανακοίνωση του 2010 είχαμε κάτι για τη στρατηγική εφαρμογής Τη χάρτα αυτή. και η Επιτροπή είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων που το επεκτείνει πέρα από τι εσωτερικέ τη πολιτικέ. Η χάρτα επίσης δηλαδή ισχύει και για την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και βάσει του άρθρου 21 ε, πρόκειται για την πρόθεση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε ολόκληρο τον κόσμο, σεβόμενοι τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και το σεβασμό όλων των αρχών που αναφέρονται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε για μια μεθοδολογία για την εφαρμογή των όσων αναφέρονται στη χαρτά. Έτσι, είχαμε την έκθεση του 2009 για την μεθοδολογία όσον αφορά το συστηματικό έλεγχο της προσαρμογής στις διατάξεις της χάρτας. Η μεθοδολογία αυτή βέβαια έχει να κάνει με τις εσωτερικές πράξεις, την εσωτερική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει οθετηθεί ακόμα μεθοδολογία όσον αφορά την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιδών Δικαιωμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βέβαια πολλές εξωτερικές δράσεις όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί η χάρτα και η δικιά μας η υπηρεσία ασχολείται για να δει ποια θα ήταν η καταλληλότερη μεθοδολογία για να εφαρμοστεί η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εργασίες της η υπηρεσία μας λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων και το έργο της Γενικής Διεύθυνσης Αγορών. Τώρα, όσον αφορά τις εγγύσεις, η χάρτα μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο και να μπορούμε βάσει αυτού να εκτιμούμε την τήρηση ή όχι των αρχών. Αλλά βέβαια χρειάζεται και συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών και να διασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρώνει τη δουλειά που γίνεται στον ΩΣΑ. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση εννοείται ότι θέλει να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Έχουμε και την κυρία Όντρε Ρόχναντ εδώ, που είναι επίση εμπειρογνώμων από την Διεθνή Αμνηστία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα κοιτάξω να περιοριστώ στα 10 λεπτά για να υπάρχει και χρόνος για ερωτήσεις. Τα σχόλιά μου έχουν ε, να κάνουν και με επιχειρήσεις αλλά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και βέβαια οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. Η εμπειρία μας στη Διεθνή Αμνηστία μετά από την έρευνα που έχουμε κάνει για τους διαφορούς φορείς που μπλέκονται τα τελευταία 10 χρόνια είναι πρακτικού χαρακτήρα προσεγγίσεις για τις ε, μη οικονομικές ε, δραστηριότητες. Έχουν αναπτυχθεί πολλές μεθοδολογίες. Όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα ή για οικονομική ενίσχυση φορέων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιος είναι ο αρνητικός αντίκτυπος τέτοιων δράσεων και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μην θέλουν οι δραστηριότητές τους να συνεισφέρουν σε παραβίαση ε, ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Αυτό είναι το βασικό για μας. Η δέση επιμέλεια είναι αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε να τηρείται και από τις επιχειρήσεις και από όσους στηρίζουν οικονομικά τις επιχειρήσεις. Να έχουν υπόψη τους τους κινδύνους και να λαμβάνουν δράσεις για να αποφεύγονται ή για να μετριάζονται οι επιπτώσεις τους. Εάν βασιζόμαστε λοιπόν στη δέσο επιμέλεια, τίθεται και διάφορα ε, θέματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κάποια πολιτική κατάλληλη για την δέουσα αυτή επιμέλεια. Τι πολιτική είναι αυτή και πώς εφαρμόζεται και ποιες είναι οι επιπτώσεις της. Όσον αφορά τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, τη δέσο επιμέλεια τη βλέπουμε είτε όσον αφορά τον ίδιο τον οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων, αλλά και όσον αφορά την επιχείρηση που υποφελείται. Η πρώτη περίπτωση σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσει στι οποίε πηγαίνει η στήριξή του οι ίδιε έχουν ένα σύστημα δέουσα επιμέλεια, προκειμένου να αποφεύγονται παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβιάσει όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Η αναφορά αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα αποτελέσματα, δηλαδή πρέπει να εντοπίζει τους κινδύνους και να βλέπει πώς αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι αυτοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αφήνεται θελοντικά στα χέρια των επιχειρήσεων, πρέπει να είναι κάτι υποχρεωτικό. Και για να λειτουργήσει αυτό στην πράξη, εμείς έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αποτελεί αυτό ένα θέμα ανατομέα. Δηλαδή, πολύ συγκεκριμένα να λέμε ότι κάθε φορά πρέπει να εξετάζεται το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το θέμα τη προστασία του περιβάλλοντο. Στι εξορρυκτικέ εταιρείε, για παράδειγμα, δεν περιμένετε βέβαια να μην γνωρίζει η εταιρεία τι επιπτώσει θα έχει η εξορρυκτική δραστηριότητα στην περιοχή και στον κόσμο. Μπορεί να υπάρξει ρήπανση από την εξόρυξη, μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα ασφάλειας επίσης. Θα ήταν προτιμότερο λοιπόν αυτό το non-financial reporting να γίνεται σε συνεργασία ε, κάθε φορά με την συγκεκριμένη επιχείρηση και τους συγκεκριμένους ειδικούς και όχι να καλύπτει όλους τους τομείς. Δύο θέματα προκύπτουν. Το ένα έχει να κάνει με την αλυσίδα ε, προμήθειας. Η όπου βλέπουμε ποιε είναι οι σε ολόκληρη την αλυσίδα στη συνέχεια. Υπάρχουν κατευθυντήριε γραμμές για το πόσο μπορεί να εφαρμοστεί η ιδέουσα επιμέλεια. Το άλλο θέμα το οποίο συχνά προκύπτει όσον αφορά τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων είναι αν αυτές δίνονται σε ε, μια επιχείρηση η οποία ας πούμε έχει αναλάβει ένα τεράστιο έργο, ένα τεράστιο φράγμα Πώς ελέγχεται τότε. Η δέσο επιμέλεια ε, σημαίνει ότι οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να φροντίσουν ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν διασφαλίσει ότι το έργο το οποίο κάνουν με την στήριξή τους δεν ελοχεύει κινδύνους ή ότι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται. Οι επιχειρήσεις όμως πολύ συχνά δεν το κάνουν παρά μόνο αν τους ζητηθεί Υπάρχουν βέβαια διαφορετικά επίπεδα δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων και πρέπει να αναφέρονται ρητά με συγκεκριμένα κριτήρια για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων. Το non-financial reporting όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια και οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να αναφέρουν και τα μέτρα μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων. Και να ξέρουμε τι βγαίνει από εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ε, περιπτώσεων που αυτό δεν γίνεται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανακαλύψουμε και πάλι τον τροχό. Αν έχουμε ένα μεγάλο σχέδιο στην Αφρική και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στο περιβάλλον, για παράδειγμα, τότε πρώτα πρέπει να ρωτήσετε τι κομμάτι γης θα καλυφθεί για το έργο αυτό, ποιοι ζουν εκεί, ε, να φροντίσουμε να δούμε ποια είναι οι εθνικές προδιαγραφές, αν θα υπάρξουν κάποια θύματα. Είναι πράγματα τα οποία έτσι καλώς υπάρχουν, δεν χρειάζεται να τα ανακαλύψουμε σήμερα. Τέλος, αν υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που δεν είναι συνήθιστοι του τομέα, αλλά κάπως έκτακτοι, τότε θέλουμε να σημειωθούν ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που ελοχεύουν και που και τους οποίους τους έχουμε συναντήσει πολλές φορές. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι η επιχείρηση θα πει. Θα πει όχι, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό το πρόγραμμα. Όμως ψάξτε το στο Google και θα δείτε ότι μη κυβερνητικέ οργανώσεις τις περισσότερες φορές έχουν επανειλημμένα εκφράσει διαμαρτυρίες και ενστάσεις για τέτοιου είδου προγράμματα. Είτε πρόκειται για το περιβάλλον, είτε πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να πει η επιχείρηση ότι δεν συμφωνεί ή ότι έχει αντεπιχειρήματα. Ακόμα δηλαδή και αν ισχύει αυτό, η προσφυγή πρέπει να γίνει, πρέπει να αναφερθούν οι κίνδυνοι. Το στοιχείο κλειδί τώρα είναι ποιες ερωτήσεις ε, θέτουμε για την αναφορά αυτή των ε, επιπτώσεων. Και πάλι εδώ πρέπει να τηρείται η διαδικασία της δέουσας επιμέλειας και να ρωτάμε τι πολιτικές ισχύουν, τι διαδικασίες ισχύουν με τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, ποιες είναι οι προδιαγραφές που εφαρμόζουν, ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές, πώς εφαρμόζονται, ποια κύρια θέματα έχουν αναφερθεί στην περίοδο αναφοράς και πώς αντιμετωπίστηκαν. Πρέπει να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη ουσιαστική έκθεση έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει πάντα και ίχνος αυτών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Οι ευρωβουλευτές τώρα έχουν το λόγο για να ρωτήσουν. Ο κύριος ε, Μορφή είναι πρώτος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση σας. Ε, διαβάζοντας το έγγραφο εργασίας ε, και την ετήσια έκθεση για τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων, επιβεβαιώνονται οι φόβοι που εκφράστηκαν στην τελευταία συνάντηση, γιατί αυτό που διαβλέπουμε είναι ότι η υποβολή εκθέσεων από τα κράτη-μέλη είναι ανομοιόμορφη. Τα περισσότερα κράτη-μέλη από τη είδα έχουν ακολουθήσει μια άσκηση τσεκαρίσματος ουσιαστικά επιλογών ενώ άλλοι οργανισμοί έχουν αναπτύξει συγκεκριμένα μέσα. Τρεις μόνο χώρες έχουν πάει πολύ πιο πέρα από τη βασική μορφή όπου τσεκάρουν ένα τετραγωνίδιο και απλά προχωράνε παρακάτω. Αυτό αναδεικνύει τα προβλήματα όσον αφορά τι απαιτήσει υποβολή εκθέσεων μέχρι στιγμή, ότι είναι ανεπαρκή οι εκθέσει και όχι επαρκώ λεπτομερεί όσον αφορά τι ερωτήσει που τίθενται και αυτό αποτυπώνει και τα προβλήματα που αφορούν τι κοινέ προσεγγίσει του ΩΣΑ. δεν αντικατοπτρίζουν ούτε καν δεδηλωμένα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Και φυσικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι νομικός δεσμευτικά. Τώρα αναφερόμενο στα θέματα του ομιλήτρες στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, δεν θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ένα μηχανισμό ώστε να εφαρμόζουμε όλα αυτά στην εξωτερική δράση. ώστε όχι απλά να αντικαταστήσουμε τις κοινέ προσεγγίσεις, αλλά να θέσουμε ορόσημα βάσει των οποίων θα αξιολογούνται οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων. Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι κατά πόσο το Συμβούλιο, η ομάδα οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων θα ήθελε να παρέμβει, όχι. Γενική Διεύθυνση Trade της Επιτροπής, κάποια αντίδραση, ναι. Ο κύριος Σόλτς. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά την πρακτική υλοποίηση του κανονισμού 1233 του 2011, αλλά εκτιμάμε το γεγονός ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι εδώ, όπως φαίνεται, συμφωνούν ότι προσπαθούμε η υλοποίηση να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. πολύ ενδιαφέρουσε οι απόψεις που ακούσαμε των εμπειρογνωμόνων και οι παρουσιάσει τους. Κατά την απόψή μα, αυτό που θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τις περαιτέρω συζητήσεις και την υλοποίηση ουσιαστικά του κανονισμού αυτού είναι επίσης ε, ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση κοινή κοινή λογική. Θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσει, αλλά αυτό να μην αποτελεί γραφειοκρατικό φόρτο για την αρχή αναφορά. Όχι να παρέχουν πληροφορίε που δεν βοηθούν του όσου θα διαβάσουν τι εκθέσει αυτέ. Επίση, πρέπει να έχουμε υπόψη μα τι είναι εφικτό όσον αφορά τους οργανισμούς υλοποίηση και να τους παρέχουμε εύλογη ευελιξία στην επιλογή του τρόπου υποβολής αναφορών εκθέσεων και επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε τα όσα γίνονται ή έχουν ήδη γίνει στον ΩΣΑ ή σε παρόμοιους οργανισμούς που και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μόνο αυτά, αλλά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως πρόταση μια αναφοράς. Τέλος, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η Επιτροπή μόλις κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος ε, της έκθεσης ε, για τις εξαγωγές. Ε, εάν υπάρχουν ερωτήσεις για αυτό το κομμάτι, ευχαριστώ να τις απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Καθώς οι εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης ε, αναφέρθηκαν απευθείας, θα θέλετε να αντιδράσετε στις, στα σχόλια. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος βουλευτής ο ΣΑ, το έγγραφο του ΣΑ, φυσικά υιοθετεί μια ευρεία προσέγγιση φυσικά δεν προσπαθούμε να την αμφισβητήσουμε αλλά η μεθοδολογία ανάπτυξης βάση του χάρτη θα μπορούσε να συμπληρώσει όσα υπάρχουν στο έγγραφο του ΩΣΑ ε, βοηθώντας να αναπτυχθεί μια πιο λεπτομερής μεθοδολογία βάσει της οποίας ε, οι εγγύησει εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούσαν να αξιολογηθούν ω προ τη συμμόρφωση. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα. Ε, για τους οργανισμούς υποβολής εκθέσεων έχει νόημα να υπάρχουν υπερβολικές και κοινωνικές προφορίες στο ίδιο επίπεδο με τις οικονομικές προφορίες, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικές για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και τη συμβολή τη. Ε, στους μακροπρόθεσμους στόχους για το περιβάλλον και στην κοινωνική της σημασία. Ε, κύριος Γιάννη Ξαντώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπενιαμπάν, τον κύριο Κίν και την κυρία Κόργαν. Πιστεύω ότι τα όσα μας είπαν είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και θα τροφοδοτήσουν την έκθεσή μας σε αυτή την Επιτροπή. Εγώ θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω αυτές τις πληροφορίες στο μέγιστο. Για άλλη μια φορά, όπως βλέπουμε, είναι ένα οριζόντιο ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό, πιστεύω, σήμερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την εξωτερική της εικόνα και για την τήρηση των στόχων της συνθήκης της. Ήθελα να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, ευχαριστώ εσάς κύριε Πρόεδρε που επιτρέψατε να πάρουμε λίγο παραπάνω χρόνο και ευχαριστώ πολύ και τους Διερμηνείς. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ε, ευχαριστούμε που ήρθατε να συζητήσετε μαζί μας ε, ε, εδώ Ολοκληρώνεται η συνάντησή μας 24 Απριλίου η επόμενη 25 η τακτική μας συνάντηση σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Sorry,